Μία ανακοίνωση όσον αφορά την απόφαση διαφόρων επιτροπών να ξεκινήσουν οι διαθεσμικέ διαπραγματεύσει με εφαρμογή του άρθρου 69.4, παράγραφο 1, που αναγγέλθηκε, αναγγέλθηκε στην ε, συνεδρίαση τη Δευτέρα. Ζήτησα αιτήματα ψηφοφορία με βάση το άρθρο 69 σε παράγραφο 2 από τι ομάδε Γκουέντζιελ, ALDE, EFTD και ECR για την απόφαση τη Επιτροπή ΚΙΛΤ να ξεκινήσουν οι οργανικέ διαπραγματεύσει με βάση τι έκθεσει για τι ε, οπτικοακουστικέ υπηρεσίε για την αλλαγή της πραγματικότητας αγοράς είναι η έκθεση Φερχάιεν Κάμερετ. Η ψήφιση, η ψηφοφορία για την απόφαση της Κίλτ να ξεκινήσουν οι οργανικές διαπραγματεύσεις θα γίνει αύριο. Όσον αφορά τι αποφάσει των επιτροπών ΙΝΤΑ, ΙΤΡΕ, ΙΜΚΟ, ΠΕΣ και ΛΥΜΠΕ για να ξεκινήσουν οι οργανικές διαπραγματεύσει, δεν έλαβα κανένα αίτημα ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο. Αυτέ οι επιτροπέ μπορούν λοιπόν να ξεκινήσουν τι διαπραγματεύσει.